Uh, uh, Καλώς. Έλεγα λοιπόν ότι έχω δύο αιτήματα. Έναν απευθύνω στους διερμηνείς, αν μπορούν να παραμείνουν για λίγα περισσότερα λεπτά για να μας βοηθήσουν. Και δεύτερον, απευθύνομαι στους κοιόδης εισηγητές να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομοι. Η συγγήτρια του άλλως είπε ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις και υποδείξεις. Κύριε Σαλαφράγκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. Να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Σαντιάγο Φίσας, ο οποίος είναι ο σκιώδης εισηγητής της πολιτικής μου ομάδας. Δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Σας συγχαίρει για την εργασία σας ελπίζει ότι οι τροπολογίες που θα υποβάλει κινούνται προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε. Θα παρουσιάσει τροπολογίες για την ενίσχυση της εμπορικής διάστασης της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής ε, αναφέροντας συγκεκριμένα εργαλεία όπως το Aid for Trade και θέλει να επαναλάβει ότι είναι διαθέσιμος να συμπληρώσει, να συμβάλλει ε, στην ε, ε, γνωμοδότηση που θα εμπλουτίσει την έκθεση του κυρίου Μωρίς Πόγκα στην αρμόδια επιτροπή ΝΤΕΒΕ. Σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε το παν για να είναι η συνεισφορά μας θετική. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος για το ECR, η κυρία Μακλάρκιν, ευχαριστώ. Ε, μιλώ εκ μέρου του κυρίου Ζαραντήλ που έχει πάρα πολύ μακροσκελή σχόλια να υποβάλει. Ω ECR, ω συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ, σα ακολουθούμε και προσυπογράφουμε διάφορε συστάσει που έχετε συντάξει κυρία Αρένα και θέλουμε ο ιδιωτικό τομέα να εμπλιακεί περαιτέρω και να εξαταστούν και άλλα προγράμματα που θα κινητοποιήσουν τοπικού χρηματοπιστωτικού και χρηματοοικονομικού πόρου για να έχουν περισσότερε δυνατότητε οι χώρε αυτέ. Όσο αναπτύσσονται, να απομακρύνονται από τους παραδοσιακούς τομείς ε, και να είναι πιο παραγωγική η γεωργία τους. Τα υπόλοιπα σχόλια θα σας τα υποβάλω, θα τα δώσω και στους κοιόδης εισηγητές, αλλά και εμείς θα συνεργαστούμε με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Στρέφομαι τώρα στην, στο Άλντε, η κυρία Λαλόν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Χαίρομαι διότι έχω την ευκαιρία να εκφραστώ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Μια σχέση εξαιρετικά σημαντική, από την οποία εξαρτάται η σταθερότητα και η ευημερία αμφότερων των υπήρων. Χαιρετίζω ε, το ε, δουλειά του εισηγητή της Επιτροπής ΝΤΕΒΕ, Μωρίς Πονκά αντοχή, η ανθεκτικότητα των αφρικανικών χωρών θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των μελημάτων μας. Θα πρέπει πράγματι να δουλέψουμε έτσι ώστε οι χώρες αυτές να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους και θα στηρίξουμε την ε, κυρία Αρένα στην γνωμοδότησή της. Θα υποβάλλουμε τροπολογίες ε, προκειμένου να ε, εμπλουτίσουμε τη γνωμοδότηση προσπαθώντας να δώσουμε απάντηση στο εξής ερώτημα. Πώς το εμπόριο θα ωφελήσει την Αφρική και θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Το εμπόριο είναι παράγοντας ανάπτυξης, αλλά ε, εμπόριο και ανάπτυξη δεν συμβαδίζουν πάντοτε. Είναι οι χώρες αυτές ε, ευάλωτες ε, ως προς τις διακοιμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών στο παγκόσμιο εμπόριο χρειάζεται να ενισχυθεί ο τριτογενής τομέας των υπηρεσιών στην Αφρικανική Ήπειρο, ε, καθώς και να ενισχυθούν οι, ε, ο δευτερογενής τομέας και το εμπόριο, και όχι μόνο η πρόταση ύλη. Το εργαλείο Aid for Trade θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Χρειάζονται αφρικανικές λύσεις στο αφρικανικό πρόβλημα. Άρα, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρθρώνεται γύρω από το σχέδιο της ελεύθερης οικονομικής ζώνης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να χρηματοδοτηθούν προγράμματα για εφόρα ανάπτυξη και για δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Αφρικανική Ήπειρο. Α σκεφτούμε την ψηφιακή αγορά, τι καθαρέ μορφέ ενέργεια, στον εξηλεκτρισμό, στον εξυγχρονισμό των υποδομών και κυρίω των υποδομών υγεία. Να στηρίξουμε την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, τον ιδιωτικό τομέα οι θύνοντες πρέπει να έχουν περισσότερες επαφές μεταξύ τους, καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, να γίνονται σύνοδοι κορυφής, όχι μόνο μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και εκπροσώπων επιχειρηματικών φορέων, εκπροσώπων ε, του, ε, ε, του ιδιωτικού τομέα το Φόρουμ των Γυναικών, των Αφρικανών Γυναικών, οι οποίες επιδεικνύουν πνεύμα επιχειρηματικότητας πραγματικά αξιοθαύμαστο, είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η πρώτη Σύνοδος Αφρικής Γαλλίας είχε ε, αφιερωθεί στις ε, Αφρικανές γυναίκες επιχειρηματίες. Εγώ παρέστην, είχα εκπληκτικές συναντήσεις με ανθρώπους, με γυναίκες εκπληκτικές και πραγματικά πρέπει να ακουστεί η φωνή τους. Γιατί έχουν πολλά αξιόλογα να πούν. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι για άλλη μια φορά. Ο κύριος Σόλτς για την ΚΟΕ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι εξαιρετικά σύντομος γιατί η σκιώδη εισηγήτρια δεν είναι εδώ, αλλά μου ζήτησε να πω ότι την άποψη της εισηγήτριας και επαναλαμβάνει ότι η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχύει το δίκαιο εμπόριο και την αλληλέγγυα οικονομία. Να μην συμβάλλει άμεσα ή έμεσα στην διαφθορά και στην φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή, να συμβάλλει στη καλή χρηστή διακυβέρνηση, στην λογοδοσία, να έχουμε ρήτρε δέουσας επιμέλειας σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες, ρήτρε για την βιωσιμότητα του χρέους των χωρών, ε, προγράμματα που δεν θα αυξάνουν το δημόσιο ε, χρέος των χωρών σε σημείο που να καθίσταται μη βιώσιμο. Θα ε, σταθώ κάπου εδώ και τα λοιπά θα τα υποβάλω αρμοδίω στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Η κυρία Χαουτάλα για τους πράσινους. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, όλοι λένε για μένα ότι δεν μακρηγορώ. Τώρα θα σας το αποδείξω για άλλη μια φορά. Πολλά από τα θέματα που θίγει η κυρία Αρένα στο σχέδιο γνωμοδότησής της είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι μπορούμε να τα αναπτύξουμε λίγο περισσότερο. Κάποια πολύ σημαντικά για εμάς. Για παράδειγμα, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος είναι στοιχείο κλειδί και αυτό έχει να κάνει με τη χρηστή διακυβέρνηση, την διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και θέλω να προτείνω κάτι πιο συγκεκριμένο ως διατύπωση για όλα αυτά. Εκτιμώ αυτό που είπε η προηγούμενη ομιλήτρια για τις γυναίκες και το εμπόριο. Εξαιρετικά σημαντικό και αυτό θα το αναπτύξουμε περισσότερο στη γνωμοδότησή μας. Και τέλος, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αηφόρο Ανάπτυξη, που είναι ακριβώς ο κατάλληλος τρόπος να εμπλακεί ο ιδιωτικός τομέας, να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη, να πούμε δύο λόγια για όλο αυτό το θέμα στην γνωμοδότηση και έτσι πιστεύω ότι θα συμβάλλουμε στο έργο της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Ευχαριστώ ε, κυρία Μπεγκίν για το EFTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τη συνάλφου κυρία Ρένα για την πάρα πολύ καλή δουλειά της. Ε, προφανώς ε, και συμφωνούμε μαζί της ε, με την προσέγγιση της. Βεβαίως και εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε να συνεισφέρουμε που σημαίνει ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα της Αφρικής. Μια Αφρική που για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζαμε ως τράπεζα και σήμερα ε, υπάρχει πλέον μια ευκαιρία για τους Αφρικανούς αλλά και για μας. Ε, κατόπιν τούτου προφανώς ε, και υπάρχει ένα κίνητρο να εξορθολογήσουμε τις εμπορικές σχέσεις ακριβώς όπως έχει γίνει και με τα ορυκτά, τις ορυκτές πρώτες Θεωρώ ότι φέρουμε ευθύνη εναντί της ε, Αφρικής, ε, όχι ψώντας τον δάκτυλο, αλλά με ίσους όρους να συνεργαστούμε γιατί είναι σημαντικό να αναλυθούν πρωτοβουλίες. Επίσης θα φέρουν πλούτο σε αυτή την ε, Ήπειρο και μην ξεχνάμε ότι στο μέλλον ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξη θα προέρχεται από την Αφρική, άρα δηλαδή το να υπάρχει σταθερότητα στην Ήπειρο αυτή είναι σημαντικό για όλους. Ο κύριος Μάρτιν ζήτησε το λόγο. Ε, πάρα πολύ σύντομος ε, θα είμαι. Παράγραφος C, κάτι πολύ μικρό. Αυτό το βρίσκω αρκετά επικίνδυνο. Λέει ότι οι ρυθμίσεις εμπορικών προτιμήσεων δεν έχουν συνεισφέρει καθόλου στο να υπάρχει σταθεροποίηση αυτή τη χώρα. Ε, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Έχουμε προγράμματα τα οποία βοήθησαν τις αφρικανικές χώρες. Αν ο στόχος σας είναι να πείτε ότι δεν αρκεί, εντάξει, αυτό σας στηρίζω. Και συμφωνώ και με άλλους αντέλφους ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για το εμπόριο, ε, να εξαλείψουμε φραγμού στο εμπόριο και όλα τα άλλα που ελέγξαν. Δεν έχουμε χρόνο, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά ξέρετε, αυτή είναι εδώ τη διατύπωση. Ειλικρινά πρέπει να την αλλάξουμε. Πρόεδρο πολύ ωραία. Και τώρα στην ε, Επιτροπή για την πιο σύντομη δυνατή παρουσίαση που μπορεί να υπάρξει ποτέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας καλέσατε να συμμετάσχουμε σε αυτό το διάλογο. Η βάση μας είναι η ανακοίνωση που έχουμε εκδώσει, αλλά όπως πάντα σε τέτοιου ανακοινώσεις πρέπει κανείς να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Τούτου λεχθέντος. Ελπίζω ότι καταφέραμε να καταστήσουμε πρώτη προτεραιότητα να δημιουργηθούν θέσει απασχόλησης στην Αφρική. Οπότε σημείο θετηρία του προβληματισμού μας ήταν το μέγεθος των δημογραφικών τάσεων στην Αφρική. Σε σύγκριση με το ρεκόρ δημιουργία θέσεων εργασία τα τελευταία δέκα χρόνια είχαν μια αναδείκτη ανάπτυξη περίπου 5% τα τελευταία 10 χρόνια με 3 εκατομμύρια θέσεις εργασία. Μέχρι το 2035 χρειαζόμαστε 15 εκατομμύρια θέσεις εργασία το χρόνο. Οπότε αυτό είναι και ο μεγάλος κίνδυνος. Ένας τρόπος να βοηθήσουμε είναι οι επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων, το EIP. Είναι η απάντηση για να δημιουργηθούν όλες αυτές τις Να εκβιομηχανίσουμε, να δημιουργήσουμε προσθέμενη αξία, λυσίδες αξίας. Ε, αυτές είναι οι τρεις κατευθύνσεις το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η συνδρομή για την βελτίωση των κανονιστικών πλαισίων και τρίτον βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Και θέλω να προσθέσω και το εξή. Υπάρχει μια πρωτοβουλία συμπληρωματικότητα, την οποία έχουμε προτείνει να βελτιώσουμε το επενδυτικό κλίμα. Και η πρότασή μας είναι μαζί με τους ομολόγους μας, μαζί με του εταίρου μα, να καθορίσουμε κατευθείαν για τι. Ε, ε, επενδυτικέ πολιτικέ για την επεξεργασία επενδυτικών πολιτικών. Ε, η συγκεντρία πολύ σωστά λέει ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε την Αφρική ως κάτι ενιαίο. Η Αφρική είναι 54-55 χώρες σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και αν θα πρέπει αυτές οι πολιτικές μας να ε, προσαρμοστούν στην περιοχή της Αφρικής, την μιλάμε. Η, η Σύνος Κορυφής έχει ως στόχο να λυθούν μέτρα έτσι ώστε να υιοθετηθούν κατευθείαν γραμμέ που θα δημιουργούν ένα πιο προβλέψιμο επενδυτικό κρίμα. Άρα λοιπόν η βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι αυτές οι κατευθείαν γραμμέ θα δώσουν βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια δικαίου, το κράτος δικαίου, καλή διακυβέρνηση, την εταιρική ευθύνη κλπ. Όλες αυτές οι κατευθείαν γραμμέ έχουν τις έχουμε εμπνευστεί από παρόμοιες αρχές της τη, του G20 και των χωρών ΑΚΕ. Δεν θα είναι υποχρεωτικέ εφαρμογή δεσμευτικέ, θα είναι συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρικανικής Ένωση επί συγκεκριμένων αρχών οι οποίε θα βοηθήσουν το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι ο λόγο στην Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις σας. Ε, θα ήθελα να καθισιάσω τον David Μάρτιν όταν λέμε ότι οι ε, εμπορικές προτιμήσεις δεν έχουν επιτρέψει την, τον, εκβιομηχάνηση των χωρών. Ακριβώς εννοούμε δεν ήταν επαρκής η εκβιομηχάνηση, συνεπώς θα πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα που ληφθεί, να σκεφτούμε άλλα μέτρα. Προφανώς δεν επικρίνουμε τις ε, προτιμησιακές, τις εμπορικές προτιμήσεις. Δεν ήταν επαρκής, αλλά ναι θα πρέπει ενδεχομένω να ξαναδούμε λίγο το κείμενο. Δυστυχώ, ε, είμαστε πολύ περιορισμένοι σε ό,τι αφορά το μέγεθος της γνωμοδότησης κάθε φορά και μερικές φορές ε, ε, το κείμενο δεν εκφράζει το ακριβώς που θέλει να γράψει ο συντάκτη. Ευχαριστώ πολύ όλου και ιδίω την Κομισιόν. Η, πράγματι αυτή είναι η λογική. Το εμπόριο, θα πρέπει να στήριξει την δημιουργία θέσεων το δημογραφικό πρόβλημα είναι τεράστιο στην Αφρική γιατί επηρεάζει πάρα πολύ και τη μετανάστευση. Αναφερθήκατε στην Νούγκταντ ε, και τις συστάσεις της. Πράγματι θα πρέπει να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή ανάμεσα στις δικές μας στρατηγικές και τις στρατηγικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο και στους κόλπους του ΟΗΕ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Καθώς επίσης και με τις περισσότερες από τις παρεμβάσεις που οποίες έκανε οι συνάδελφοι θα συνεργαστούμε για να συμπληρώσουμε αυτή τη μικρούλα γνωμοδότηση, ε, την ολιγοσέλιδη και ολιγόλογη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την αισιοδοξία σας. Ε, τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ θυμηθείτε ότι το περιεχόμενο